Μετά την παρέτηση της κυρίας Βίκη Μέιερ, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι χειρεύει θέση της από τις 16 Μαρτίου του 2017 και βάσει του κανονισμού ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ο κύριος Γιάζεκ